Good afternoon, colleagues. Oh. ask you to take seat, please? Καλησπέρα σας συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε για να ξεκινήσουμε. Καλωσορίσατε και πάλι στο Κοινοβούλιο μετά την θερινή διακοπή. Έχουμε πολλή δουλειά αλλά όχι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση Επιτροπής, όπου η ατζέντα δεν είναι πολύ φορτωμένη, Παρ' όλα αυτά αρχίσουμε να δουλεύουμε. Μπορώ να θεωρήσω εγκεκριμένη την ημερήσια διάταξη. Ναι. Επίσης τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Σας ευχαριστώ. Και τώρα κάποιες ανακοινώσεις από μένα. Πρώτον, για, την για τον κατεξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, τα τεχνη, για τις τεχνικές προδιαγραφές της Οδηγίας 2013-36 η οποία αναθέτει ε, αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσβαση στις δραστηριότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των ε, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίω στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 147 και των άρθρων 35, 36 και 39 και βάση του άρθρου 139 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μπορεί να φέρει αντίρρηση το Κοινοβούλιο στην έγκριση της πράξης αυτής. Ε, η προθεσμία για υποβολή των ενδεχομένων αντιρρήσεων είναι 21 Οκτωβρίου. Μία σχετική απόφαση για, τις κατεξοδότηση πράξης, για την κατεξοδότηση πράξη αυτή θα ληφθεί και στη συνεδρία των συντονιστών στις 23 Σεπτεμβρίου. Και στις 23 λύγει και η προθεσμία για οποιαδήποτε πρόταση από τον εισηγητή ή τους συναδέλφους για την ε, καταψήφιση μιας τέτοιας κατεξοδότησης πράξης. Να σας ενημερώσω για τους οικονομικούς διαλόγους επίσης μετά την συνεδρία των συντονιστών στις 22 Ιουλίου ο... η Πορτογαλίδα Υπουργό Οικονομικών κ. και συμφώνησε να συμμετάσχει στον οικονομικό διάλογο που θα διοργανώσουμε στις 2 Δεκεμβρίου ενώ ό,τι αφορά την Γαλλία και μετά την ακύρωση των γύρων οικονομικών διαλόγων έχουμε έρθει σε επαφή με, τον, με το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και σκοπεύουμε το φθινόπωρο να οργανώσουμε συζήτηση οικονομικού διαλόγου με την Γαλλία, που δεν έχει όμως οριστεί ακόμα. Τέλος, να ενημερώσω τα μέλη ότι οι συντονιστές συμφώνησαν η Επιτροπή να συνεχίσει την εργασία της σε ό,τι έχει μείνει σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη θητεία και ενημέρωσα τον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων επιτροπών αναλόγως και επίσης τον Ιούλιο και πάλι οι συντονιστές συμφώνησαν για την κατανομή των θεμάτων μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, τα ταμεία των χρηματοπιστωτικών αγορών, benchmarks για την ALDE, διαφάνεια και διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σοσιαλιστές και δημοκράτες, διαφορετικά μέτρα για την ενθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ΕΛΚ, αναδιατύπωση δραστηριοτήτων και εποπτείας των συνταξιδοτικών ταμείων ΕΛΚ, στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών το διεθνές, της Υπηρεσίας Διεθνούς Εμπορίου και τις ξένες επενδύσεις πράσινη, κανονισμός του Συμβουλίου για τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές, σύσταση για κανονισμό του Συμβουλίου για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Πρόεδρος, Γενικός Προπολογισμός 2015 Άλντε. ήδη πόροι Βάση του FTT ALDE, Κοινωνική Σύνοδος ΓΚΟΕ, e, τροποποίηση της οδηγίας 26-2007 για την ενθάρρυνση των ε, μακροπρόθεσμων μετόχων και τις οδηγίες, την αναδιατύπωση τη οδηγία 24-2003 Σοσιαλιστές και Δημοκράτε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τον Συντονισμό Πολιτικών 2014 ALDE, Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής 2014 ΕΛΚ, Ετήσια Έκθεση για τον Ανταγωνισμό 2013 2013-Συντερική και Μεταρρυθμιστέ, Ετήσια Έκθεση για τη Φορολογία Σοσιαλιστές και Δημοκράτε, οικονομική διακυβέρνηση και σχετικέ κατευθυντήριε γραμμέ σοσιαλιστέ και δημοκράτε. Uh, uh, Αυτά. Και να περάσουμε τώρα στο σημείο 4 της σημερινής διάταξης. Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015. Εισηγητής, ο κύριος Τόρφαλτς. Σας δίνω το λόγο. Sorry, Chair, I'm speaking on behalf of Mr. Uh, Πρόεδρε, συγγνώμη, θα μιλήσω εξ, εξ ονόματος του κύριου Τόρβαλτς. So, um, Mr. Torvalds cannot be here this afternoon. Ο κύριος Τόρβαλτς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα γιατί έχει και μια έκθεση την οποία καλείται να παρουσιάσει στην ε, Καθήλυνη Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα μιλήσω λοιπόν εξ ονόματος του εν συντομία. Καταρχά. ο εισηγητή θα ήθελα να επενθυμίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε έντονα την δημιουργία ε, μιας ε, Ευρωπαϊκή εποπτική αρχή και πιστεύει ότι η Ένωση θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω την εποπτεία σε κοινωτικό επίπεδο και ω εκ τούτου είναι πολύ ικανοποιημένο που οι πιο πολλές πολιτικές ομάδες συμφωνούν με την ανησυχία του σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο σημαίνει μείωση σε ό,τι αφορά την, ε, τη χρηματοδότηση του προπολογισμού των τριών θεσμικών οργάνων το 2014. Θεωρεί ότι θεσμικ, τα θεσμικά αυτό όργανα, οι αρχές αυτές είναι ακρογωνιαίος λήθος για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικλείδα ασφαλείας για την ανάκαμψη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ο εισηγητής ως εκ τούτου εξέφρασε την ελπίδα του να επανέλθουν ε, τα στοιχεία του προϋπολογισμού με την ψηφοφορία αυτή, τα αρχικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τα χρηματοδότηση των ESA ε, πιστεύει ότι οι τρέχουσες ε, διατάξεις χρηματοδότησης βασίζονται σε ένα μεικτό σύστημα που είναι άκαμπτο, γραφειοκρατικό και απειλεί την ανεξαρτησία των ESA. Συμβαστική τροπολογία που καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει ένα νέο σύστημα χρηματοδότηση μέχρι το 2017, ένα σύστημα το οποίο θα βασιστεί αποκλειστικά μόνο στην εισαγωγή τέλων από του παράγοντες τη αγορά, θα βασίζεται σε αποκλειστική χρηματοδότηση από ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού. Και τέλο, ο εισηγητή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλου του διαφορετικού ε, σκιώδει εισηγητέ για την επικοδομητική σου εργασία για την έκθεση αυτή. Sorry. Now I give the... Ο πρόεδρος. Το λόγο λοιπόν έχουν τώρα οι σκιώδεις. Να ξεκινήσουμε από το έλικα. Η Ιβάνα Μαλετίτσου. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Στόχος μας, δεδομένων των περιορισμών που μας επιβάλλει ο προϋπολογισμός, είναι να προωθήσουμε τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, της πρόοδου σε ό,τι αφορά το χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό. Όπως ε, υπογράμμισε ο εισηγητής, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι τρεις αρχές. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στις τροπολογίες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την, ε, τον προπολογισμό των τριών ε, αρχών. Θέλουμε λοιπόν να υποστηρίξουμε αύξηση του προπολογισμού. Σας καλούμε να υπερψηφίσετε την 6, 7, 2, 7, 6, 7, 2, 8, 2 και 2, 9 γιατί αν υπερψηφιστούν αυτές οι τρεις τροπολογίες, οι 6, 7, 07, 08 και 09 θα υπερψηφιστούν επίσης. Το ποσό που προτείνεται στις τρεις πρώτες τροπολογίες είναι πιο υψηλό από τις 67, 07, 08, 09 γιατί καταλαβαίνουμε ότι μετά από επικοινωνία με τις αρχές αυτές ότι λόγω αύξησης του προσωπικού σημαντική θα πρέπει να υπάρξουν περικοπές σε άλλες γραμμές και δεν θα υπάρχει πλέον περιθώριο για εκπαιδεύσει, αναλύσεις, έρευνα που είναι όλα απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία τους. Ζητούν λοιπόν αύξηση αρχές αυτές, τα οργανισμοί αυτοί, μόνο λόγω της αύξησης του προσωπικού. Είναι σημαντικό όμως να μην αυξηθεί μόνο η ποσότητα, αλλά και η ποιότητα. Άρα πιο υψηλό προπολογισμό. Αυτό ζητάμε. Επίσης, σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε και τη δεύτερη τροπολογία. Την 6715. Για ένα νέο προϋπολογισμό για την επικοινωνία. Να είμαστε κατά είμαστε κατά της ε, διαφύλαξης ε, πόρων. Γιατί? Γιατί θέλουμε καλή και γρήγορη εφαρμογή σε επίπεδο επιτροπής. Και με τη διαφύλαξη τέτοιων πόρων δεν μπορεί να κάνει τις νέες δεσμεύσεις που χρειάζεται η Επιτροπή και έτσι καθυστερείται όλη η διαδικασία. Και ο δεύτερος λόγος είναι σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Αν δεν υπάρχει σωστή λειτουργία, το πρώτο βήμα είναι πολύ καλύτερο να περιλαμβάνει ακροάσεις στο Κοινοβούλιο και να ζητείτε παρουσίαση των δραστηριοτήτων των ενέργειων και μόνο μετά, αν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα ως εργαλείο για να πείσουμε τις επιτροπές, ε, την Επιτροπή να λειτουργήσει καλύτερα. Αλλά δεν είναι καλό να ξεκινήσουμε κατευθείαν με αποθεματικό. Να καταψηφίσουμε. Προτείνω. Τέλος, να σας πω γιατί εισαγάγουμε την προφορική τροπολογία 1. Θα θέλαμε να εισαγάγουμε μία προφορική τροπολογία, να προσθεθεί το αν αποδειχτεί από την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και με τη φράση αυτή, τι θέλουμε να αποφύγουμε, να μην οριστεί μία λύση εκ των προτέρων για το σύστημα χρηματοδότησης. Γιατί θα πρέπει πρώτα να γίνει μια σοβαρή αξιολόγηση, μια ανάλυση αντικτύπου και αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις τρεις τα αυτά όργανα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει Πρόεδρος. Και τώρα να περάσουμε στο Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Λούντινγκσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα η διαδικασία, αλλά νομίζω ότι είναι καλά το τελικό κείμενο παρόλα αυτά. Σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς υποπτίας, θα πρέπει να αποστείλουμε μια σαφή εικόνα ότι το θέμα δεν μπορεί να είναι να μειώσουμε τους πόρους, δεν μπορεί να είναι υπερικοπή. Θα πρέπει να είμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενο όγκο δουλειά τα επόμενα χρόνια στο άμεσο μέλλον. Και το μοναδικό λογικό λοιπόν βήμα θα ήταν να υποστηριχθεί ποιοτικά η δουλειά. Και πώς θα γίνει αυτό με περικοπές. Για να βρούμε λοιπόν το σωστό προϋπολογισμό θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις ανάγκες σε πόρους και να δούμε λοιπόν τι ζητούν και οι ίδιες, τα ίδια τα ίδια ίδιοι οργανισμοί. Τα αριθμητικά στοιχεία που μας χορήγησαν οι αρχές αυτές φαίνεται ότι είναι αρκετά λογικές. Προφανώς και χρειάζονται πόροι για να εκτελέσουν το έργο τους. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε και το επίπεδο το οποίο προβλέπεται προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο έτος ε, για τις αρχές αυτέ, για το χρηματοδοτικό μοντέλο και πώς θα δημορφωθεί σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο πολλά, τους πιο πολλούς πόρους. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αμφιλεγόμενο. Γιατί είναι γνωστό ότι υπάρχουν δυσκολίες από πλευρά των εθνικών αρχών και υπάρχει άμεση εξάρτηση από τις εθνικές αρχές και αυτό φυσικά βάζει ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία των ευρωπαϊκών αυτών αρχών. Βλέπω λοιπόν ότι έχει διαμορφωθεί πλέον συμβιβασμό, τον οποίο και θεωρώ σωστό, προκειμένου να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μοντέλο σε ό,τι αφορά τη λειτουργία βάση των εισφορών θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ενδεχομένω και τέλεια από τους παράγοντες της αγοράς. Τέλος, να σας πω και το εξής από δικής μου πλευράς και κλείνω. Σε ό,τι αφορά τους φόρους, θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες προκειμένου να δούμε τι θα γίνει και στο πλαίσιο του 2020. Και εδώ η πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν είναι αποδεκτή σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία. Κοιτάξτε, ο τομέα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να μειώσουμε τη σημασία του. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλου του συμμετέχοντε για την θετική και επικοδομητική συνεργασία και με χαρά θα ακούσω τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Όλε, από την ομάδα ECRK. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Η ομάδα μας ε, έχει μια σαφή θέση συνολικά δηλαδή για τον προϋπολογισμό, δεν στηρίζουμε καμία αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού. Και θα πρέπει αν υπάρξει αύξηση σε ένα κονδύλι να αντισταθμιστεί αυτή από μείωση ίδιου ύψους σε ένα άλλο κονδύλιο του προϋπολογισμού. Αυτή είναι η άποψή μα. Το ανέφερε ε, στη γνωμοδότηση ο για τη χρηματοδότηση εγώ πιστεύω ότι όταν ε, δημιουργήσουμε, μάλλον όταν δημιουργήσαμε αυτούς τους εκτελεστικούς οργανισμούς, θέλαμε να εποπτεύονται από τις εθνικές αρχές, θέλαμε να υπάρχει ένα ενιαίο rule book για τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όχι όμως άμεσα να υποπτεύουν τους συμμετέχοντες στην αγορά. Άρα δεν θα πρέπει να λαμβάνω χρηματοδότηση βάσει αυτού του μοντέλου επειδή συνιστούν ένα κόστος, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν αναλόγως ε, αυτοί οι οργανισμοί. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου δεν μπορεί να στηρίξει το συμβιβασμό ή τη γενική κίνηση για αλλαγή ε, του μοντέλου του οργανισμού με, αυτό, με αυτή την πρόταση, με αυτό το συμβιβασμό που προτείνουμε. Δεν θα στηρίξουμε λοιπόν αυτό το συμβιβασμό. Thank you, Kay. Σας ευχαριστώ, Κέι. Η πράσινη, ο Σβέν. Or someone I'm a bit surprised because... Uh, Εκπλήσωμαι. Κάπως. Αναστρέψτε λίγο τη σειρά, τέλος πάντων, ε, για να είμαι ευγενικό. Βιέγκα Γκούε, συγγνώμη. Λάθος είδα τη σειρά, λέει ο πρόεδρος. Εκ της Γκούε, να επιστρέψω την φιλοφρόνηση. Ε, λείπει βέβαια ο αρμόδιος ε, εξημών. Έχουμε καταθέσει τις τροπολογίες μας και δεν έχουμε διατυπώσει κάποια άλλη παρατήρηση στην παρούσα Σβέν, δεν θα σχολιάσω κάτι άλλο. Ε, ήθελα να με ευγενής απλά. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να αναφέρουμε ότι χάρη στον εισηγητή καταλήξαμε σε συμβιβασμούς ό,τι φορά τα βασικά ζητήματα. Στηρίζουμε λοιπόν τη βασική γραμμή. Το βασικό είναι ότι αν ε, επισκεφτήκατε ποτέ αυτούς τους οργανισμούς ε, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στη Φραγκφούρτη και αν συγκρίνετε αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει και συμπεριλάβει στη νομοθεσία μας ε, Έχουμε 402 κατεξοσιοδότηση πράξης. Ε, υπάρχουν όμως ε, κάποια αιτήματα, ε, θέλουν κάποιους πόρους, είναι πολύ μετριοπαθή τα αιτήματά τους. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς νομοθετούμε και στερούμε από τους οργανισμούς αυτούς εν συνεχεία το προσωπικό που χρειάζονται. Είναι απόλυτα θεμητά τα αιτήματα των οργανισμών. Πέραν τούτου δε, πρέπει να πω ότι και από οικονομική σκοπιά το κόστος εσωτερικεύεται όπως προτείνεται στο συμβιβασμό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι οποίοι οφείλονται για το κόστος θα πρέπει να απομιστούν μέρος του κόστος. Αυτό είναι θεμητό, είναι λογικό. Στηρίζουμε όμως και τις προφορικές τροπολογίες του ΕΛΚ, δηλαδή να μην κλείσουμε ήδη την πόρτα προς την εξέβρεση λύσης. Είναι μια διατύπωση που μας βρίσκει σύμφωνος. Νομίζω ότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση κατά βάση. Συμφωνώ βέβαια ότι πάντοτε θα πρέπει να αναζητούμε και ενδεχόμενες εξοικονομήσεις πόρων. Με την ΕΦΡΑΚ και το Ευρωπαϊκό Προτύπων είχαμε συζητήσει και προτείναμε να παγώσουν οι αυξήσεις που είχαν προταθεί. Μακρά ήταν η συζήτηση που είχαμε μαζί τους, είχαμε και την έξω του κ. Στόλογιαν, δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση, το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί το πεδίο δράσης. Τώρα όμως λαμβάνουν αύξηση στον προπολισμό. Αυτό δεν το κατανοούμε. Δυστυχώς ε, δεν καταφέραμε να μας στηρίξει ο φιλελεύθερος εισηγητής για μείωση του προπολογισμού, αλλά παρόλα αυτά θα ψηφίσουμε υπέρ, γιατί μιλάμε για μετροπαθή μείωση. Πάντως, εν γέννη, όπως είπα, μας ικανοποιεί η πρόταση όσο έχει κατατεθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Σβέν. EFDD. Μάρκο Βάλι. Yes, it is possible. Ναι, γίνεται. Ευχαριστώ για, και τον εισηγητή για την υποβολή αυτών των προτάσεων που δείχνουν ποια είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των υποστηρικτών της για την ε, ρύθμιση του City στο Λονδίνο, της μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής αγοράς στην Ευρώπη και μεγάλο σημείο παραγωγής για όλη την Ευρώπη. Σε σχέση με όσα είχαμε συμφωνήσει παλιότερα στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή, είναι πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τώρα πώς τοποθετούνται οι σκιώδεις εισηγητές για την απορρίθμιση που βλέπουν να, προβλ... να τα ερχόμενα χρόνια στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι εδώ η κατεύθυνση που ακολουθούμε είναι ε, εσφαλμένη. Πρέπει να μειώσουμε την βαρύτητα αυτών των ε, ρυθμιστικών μας παρεμβάσεων, ώστε να μπορέσουν ελεύθεροι επιχειρήσεις να αναπτύσσονται. Ο δεύτερος βασικός λόγος ε, που είμαστε αντίθετοι στην έκθεση αυτή είναι το αίτημα να καταβάλλονται αντίτιμα από τους συμμετέχοντες στην αγορά. Δηλαδή πρόκειται για φορολογία από την πίσω πόρτα, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και των χρηματοπιστωτικών των θεσμικών τη οργάνων. Αυτό δεν είναι αντικείμενο συμφωνία από τη κυβέρνηση, ούτε αποτελεί περιεχόμενο συνθήκη. Οπότε δεν είναι θεμητό. Και βεβαίω ήδη φορολογούνται διπλά οι συμμετέχοντε στην αγορά, ιδιαίτερα σε χώρε όπω οι δικέ μα, με την αρμόδια οικονομική αρχή, που δεν σημαίνει ότι αν φορολογηθούν μία φορά ε, θα φορολογηθούν λιγότερο, απλώς δεν νομίζω ότι ακόμη και αν καταβάλουν φόρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν ελαφρύνσει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει αυτό. Ο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο θα είναι αρνητικό και χρηματοοικονομικέ υπηρεσίε που θα πρέπει να καλύπτουν το κόστο των ρυθμιστών του με τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ευρωπροτάσει. Ουσιαστικά διευρύνει ένα σύστημα που μα ανησυχεί. Δηλαδή και σε άλλες επιτροπές του Κοινοβουλίου, λόγω χάρη στην Επιτροπή Αλίας, τι θα τους πούμε, να προτείνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά της Αλίας να πληρώνουν τους ρυθμιστές της Αλίας ή να πληρώνουν οι Γερμανοί βιομήχανοι την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ρυθμίσεις που θα προβλέπει και θα τους αφορούν. Όλα αυτά είναι τελείως παράλογα, είναι κατά των συνθηκών και είμαστε αντίθετοι. Ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Μπούλκα Πάλτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΟΝ πριν από τις τερνές διακοπές ε, μίλησα για τον προϋπολογισμό του 2015 και άσκησα σαφή κριτική σε ό,τι αφορά την ε, χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αρκεί και πραγματικά είναι πολύ κοντόφθαλμος βρίσκω αυτά που ορίζονται ως ε, New Tasks Authority θα πρέπει να σημαίνει και κάτι αυτό για τον προϋπολογισμό. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν τα μέσα για να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και για να μπορούν να εγγυώνται το ίδιο επίπεδο ε, και την ίδια ποιότητα συνεργατών, υπαλλήλων. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ταχθούμε εμείς από πλευρά του ΕΛΚ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, μας απασχολεί πολύ. Η περικοπή του προϋπολογισμού για την επικοινωνία είναι κάτι το οποίο εμείς ως ΕΛΚ δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό επικοινωνίας για την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και για το ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό τώρα στην τρέχουσα συγκυρία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώσει για την Οικονομική Ένωση και για τις πρόοδους που έχουν σημειωθεί. Κλείνοντας, καλώς ορίζεται το γεγονός ότι τα πλατικά έργα θα αξιολογηθούν εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προϋπόθεση για τα έργα ε, σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές δράσεις, τα preparatory actions όπως ονομάζονται και είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια ποικιλία τέτοιων εμπλεκόμενων φορέων. Και στο πλαίσιο αυτό είναι καλό και το χαιρετίζουμε, το αναφέρω και το υπογραμμίζω, ότι με την ε, ερευνητική ομάδα, την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δημιουργήθηκε μια νέα τέτοια υπηρεσία και είμαι βέβαιος ότι αυτό μπορούμε να το επεκτείνουμε κι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Τζιλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές και τους κιόδες για το έργο το οποίο επιτέλεσαν στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Και εγώ θα εστιάσω στις Ευρωπαϊκές οπτικέ Αρχές. Καταρχάς αναγνωρίζω ότι είναι σημαντικοί οργανισμοί ε, ιδρύθηκαν πριν απο δυο 2-3 χρόνια και οι προπολογισμοί τους ε, καλύπτονται από συνεισφορά των εθνικών αρμόδιων αρχών κατά 60% και από τον κοινοτικό προπολογισμό κατά 40%. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πολλοί νέοι τομεί νομοθεσία, πολλά νέα νομοθετήματα εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί έτσι το χαρτοφυλάκιο αυτών των οργανισμών, αυτών των αρχών. Δεδομένου όμω του ότι είναι νέοι αυτοί οι οργανισμοί σχετικά και από ό,τι φαίνεται δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν πλήρως ε, τους προπολογισμού. τους. Μήπως θα ήταν πρόωρο και πρόημο να τους δώσουμε τώρα αυτή την αύξηση. Στρεφούμε λοιπόν προ τον εισηγητή και τον ερωτώ. Με ποια συλλογιστική, με ποια λογική προτείνεται την αύξηση, ιδίω λαμβάνοντα υπόψη ότι το καλοκαίρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 8 Αυγούστου δεσμεύτηκε και είπε ότι θα δρομολογήσει προπαρασκευαστικό έργο για τη βελτίωση των χρηματοδοτικών διευθετήσεων των ε, Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, ώστε να μπορούν να επιτελούν την εντολή τους, λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Καλό θα ήταν να περιμένουμε και μετά να λάβουμε αυτή την πολιτική απόφαση. Είμαι για 8 χρόνια μέλος Επιτροπής Υπερπολογισμών και γνωρίζω ότι με την αύξηση αυτή που προτείνει η Κομισιόν ε, δεν θα μας ε, δουν και πολυθετικά, ε, δεν θα το καταλάβουν εύκολα. Πρέπει να υπάρχει και ένας βαθμός αξιοπιστίας. Υπάρχουν και άλλα, όπως είναι τα πιλωτικά προγράμματα, τα οποία επίσης πρέπει να υποστηριχθούν. Έχω λοιπόν επιφυλάξεις για την προσέγγιση που ακολουθούμε. Και επειδή έχω υπάρξει και επιχειρηματία, σαν δεν μπορεί κάποιος να προσελκύσει τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Τι λέμε εμείς, δώστε σε αυτόν περισσότερα χρήματα ή καλύτερα να τους δώσουν περισσότερες επιλογές. Και να μείνουμε στα ανώτατα ποσά αυτά. Η Κομισιόν είναι εδώ. Ερωτώ, ποια είναι η θέση της Κομισιόν. Διάβασαν εκπρόσωποι της Κομισιόν την έκθεση του εισηγητή και έκαναν κάποιες δηλώσεις πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουν αλλάξει άποψη στο μεταξύ, από τότε δηλαδή που πρότειναν τον προπολογισμό αυτό. Ευχαριστώ, Βέρνερ Λάγκ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος το ανέφερε αυτό ότι εδώ και χρόνια προσπαθούμε να αναπτύξουμε τις δικές μας επιστημονικές ε, δυνάμεις για αντικειμενική πολιτική αξιολόγηση, προκειμένου να υπάρχει και πολιτική κατεύθυνση. Άρα βρισκόμαστε σε καλό δρόμο και δημιουργήθηκε μια τέτοια καινούργια υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τροπολογία 6713 αναφέρεται στην ε, συγκεκριμένη, στο συγκεκριμένο τίτλο. Το συζητήσαμε αυτό, μιλάμε για μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Δημιουργήθηκαν λοιπόν οι ε, υπηρεσίες αυτές με ε, μεγάλη ομοφωνία ως πλωτικό έργο, με περιορισμένη διάρκεια μέχρι το 2015 και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόταση για τον προπολογισμό έθεσε το τελευταίο συντολιστή για το 2015 και τι θα γίνει μετά το, την ε, κατάργηση. Και η τροπολογία των συναδέλφων υπό ηγεσία των πρασίνων τι ορίζει ότι θα αυξήσουμε τα μέσα τις άμεσες πληρωμές για 1,75 εκατομμύρια και το ίδιο σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις πληρωμών. Το πρόγραμμα αυτό τι σημαίνει ότι θα πάυσει το πρωτικό πρόγραμμα, αλλά στο τέλος το έτος 2015 θα έχουν 17,5% των ε, της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκές πηγές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μεμονωμένο τέτοιο όργανο από εθνικά κράτη-μέλη και ότι τα θεσμικά όργανα τα οποία αναφέρονται στην ετήσια έκθεση και παρά το γεγονός ότι στην αιτιολογία αναφέρεται ότι Τα μέσα αυτά χρησιμοποιούνται για δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλυφθεί και επειδή χρειαζόμαστε λοιπόν, όπως έχουμε πει, ε, δικές μας δυνάμεις, γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά της αύξησης των μέσων τέτοιων υπηρεσιών που δεν είναι αντικειμενικές. Και αυτό το λέω ενδεχομένως να χάσουμε στην ψηφοφορία. Αλλά, σήμερα, αλλά θα προσπαθήσω μέσω τη Επιτροπή Προπολογισμού και του κυρίου Λαμασούρ να προωθήσω αυτό το επιχείρημα στο Κοινοβούλιο. Γιατί στι διάφορου προπολογισμού θα, κάνουμε, θα ξεκονομήσουμε εκατομμύρια ε, ολόκληρα. Και τώρα να δώσουμε σε αυτή τον οργανισμό μία εγγύηση τη χρηματοδότηση δεν είναι δυνατόν. κύριος Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 6706, την οποία έχω καταθέσει και η οποία αφορά την χρηματοδότηση των νησιών του Αιγαίου. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, εδώ η χρηματοδότηση μειώνεται κατά 99%. Δηλαδή, ενώ υπήρχε ένα πρόγραμμα επιτυχημένο, το πρόγραμμα POSEI, για τα νησιά του Αιγαίου και πέρυσι η πρόβλεψη ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ και, το και την προηγούμενη χρονιά για το 2003 η εκτέλεση του προϋπολογισμού δείχνει ότι αξιοποιήθηκαν αυτά τα κονδύλια και πράγματι χρηματοδοτήθηκαν επενδύσεις της τάξης των 16 εκατομμυρίων, τώρα ξαφνικά εξαφανίζεται αυτό το ποσό και δεν υπάρχει. Σε μια φάση που όπως έχει δεχθεί και αυτή η Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο το μνημόνιο με την πολιτική του και την πολιτική της τρόικας φτωχοποίησε την ελλάδα μείωσε το αεπ κατά. 25%. ζητούμε λοιπόν να επανέλθει αυτό το ποσό δηλαδή να προσθεθούν 17,800 εκατομμύρια ευρώ και να έχουμε πάλι το ίδιο ποσό για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που ενισχύει τα μικρά νησιά του Αιγαίου, ένα πρόγραμμα που βοηθά στη μεταποίηση, βοηθά στη στήριξη των αγροτών, στη στήριξη των κτηνοτρόφων. Με αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσουν τα χιλιάδες μικρά νησιά του Αιγαίου τη δικιά τους οικονομική ζωή, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν, θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Θα μπορέσει έτσι να ενισχυθεί ο κανονικός εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου με βασικά προϊόντα. Αυτή λοιπόν την πρόταση έχω καταθέσει ως τροπολογία. Ζητώ από την Επιτροπή σας να την εγκρίνει για να μπορέσουν τα μικρά νησιά του Αιγαίου και οι κάτοικοί τους να αντεπεξέλθουν στις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που δημιούργησε η μνημονιακή πολιτική της Τρόικας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνω το κατάλογο των ομιλητών. και ο Σβέν Κίγκολτ ε, θα επανέλθει πολύ σύντομα. Κυρία Μπερές, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε αυτή τη συζήτηση που μας επιτρέπει να θέσουμε σε ισχύ κάποια αποπτικά εργαλεία για, την επόμενη, για τις επόμενες κυρίως χρονιές. Όπως είπε και ο συνάδελφος Όλε, στηρίζω και εγώ την πρόταση να έχουμε έναν προϋπολογισμό για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που να είναι ισοδύναμος με αυτό τον οποίο οι ίδιες θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη η χρονική περίοδος για τους οργανισμούς αυτούς και παρά της ε, δημοσιονομικές αυστηρότητας ή λιτότητας, για αυτές τις εποπτικές αρχές γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό τις χρειαζόμαστε και πόσο σημαντικό είναι να τις περικοδοτήσουμε με ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους που θα τους επιτρέπουν να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά τους. Τα προηγούμενα χρόνια ίσω είναι από του λίγου τομεί αυτό, όταν επισημιώσαμε πρόοδο. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτέ τι αρχέ να του δείξουμε ότι θέλουμε στο Κοινοβούλιο να τι ενισχύσουμε. Το έχουμε άλλωστε κάνει σε όλη τη διάρκεια τη προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδου. Αυτή είναι η αρχή που μα διέπει οι σοσιαλιστέ τώρα. Για το ΕΦΡΑΚ δεν πρόκειται για εποπτική αρχή, είναι μια δομή η οποία έχει να κάνει με τη λογιστική τυποποίηση. Έγινε ένας ε, υπολογισμός από τον προηγο... ένας απολογισμός από τον κύριο Μέστατ στην προηγούμενη ε, θητεία του Ελληνικού Συνεδρίου. Είναι πολύ αναλυτικός απολογισμός και νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τις προτάσεις ε, των πρασίνων και προς το παρόν να μειώσουμε το κονδύλι της δομής αυτής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Finance Watch, με ένα πιλωτικό σχέδιο ουσιαστικά τι δυνατότητα υπάρχει να ξεκινήσει μια διαδικασία που φαίνεται να είναι μακρόπνοη. Εγώ ποτέ δεν είδα σε καμία συζήτηση να ξεκινώνουν με αυτόν τον τρόπο πρωτοβουλίες ε, θνησιγενείς. Δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά πρέπει να ξεκινάμε κάτι, να μελετάμε τη σκοπιμότητα και τη, την, ε, το, το, εφικτό του και έπειτα να δούμε κατά πόσον αυτό θα ισχύσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ήμουν ε, κατά έναν τρόπο ανάδοχος του Finance Watch, και αυτό και δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη λογική του κ. Λάγκεν για τη δομή αυτή που είναι πολύ απαραίτητη, ιδίως εφόσον όλοι ανησυχούμε για την κατάσταση των κυβερνητικών οργανισμών και όλων όσων δεν ανήκουν στον οικονομικό κόσμο και δεν αντιπροσωπεύονται στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο. Very quick. Ευχαριστώ πολύ. Σβέν πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα μόνο να πω εν συντομία το εξής. αυτή η αντιμαχία γίνεται σιγά σιγά παράδοση στο Κοινοβούλιο. Αλλά το βασικό θέμα φυσικά δεν είναι να δημιουργηθεί ένας επιπλέον ουδέτερος παράγοντος, αλλά να κοιτάξουμε τα 300 εκατομμύρια ανά έτος που δαπανώνται σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό κάθε έτος. Ε, μία μικρή διόρθωση λοιπόν ε, αυτής της ανισορροπίας. Το γεγονός ότι δημιουργούνται ήδη οι πόροι του Κοινοβουλίου, μια μικρη διορθωση λοιπον αυτης της ανισορροπιας το γεγονος οτι δημιουργουνται ηδη οι ποροι του κοινοβουλιου ενταξει αυτο ειναι σωστο αλλα οχι αλλο μια οργανωση και ήθελα να πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τάχθηκε υπέρ ε, A-rating αξιολόγησης τέτοιας του οργανισμού αυτού. Και έτσι λοιπόν Αναφέρομαι σε αυτό που είπε ο κ. σε σχέση με την διαγραφή των, ε, της χρηματοδότησης αυτής. Ευχαριστώ να δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα σύντομα σχόλια. Πρώτα απ' όλα για τις υποπτικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη των περισσότερων μελών για τη σημασία, την καθοριστική σημασία των εποπτικών αρχών. Πρέπει να χρηματοδοτούνται σωστά. Η πρόταση της Επιτροπής, όπως ξέρετε, φέτος βασίζεται, βασίζεται στο να παραμείνουμε πιστοί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τα συζητήσαμε και στις 27 Ιουλίου. Ωστόσο, ξέρουμε ότι υπάρχουν και κάποιες αποκλήσεις της απόψης στην Επιτροπή εδώ για την αύξηση των πόρων στον προπολογισμό του 2015 το οποίο θα επηρεάσει όλη τη διαδικασία του προπολογισμού βέβαια. Σε ό,τι αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση των εποπτικών αρχών, αναφέρθηκε αυτό. Η αναθεώρηση της λειτουργίας των εποπτικών αρχών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναφέρει και η θέση μας παραμένει η ίδια. Θα εξετάσουμε τις προποθέσεις χρηματοδότησης των εποπτικών αρχών για να ληφθούν υπόψη και οι νέοι δημοσιονομικοί περιορισμοί. Κάποιες από τις παρατηρήσεις που έγιναν εδώ θα ληφθούν υπόψη όταν δούμε τη χρηματοδότηση των αρχών στο μέλλον. λόγω χάρη την εξισορρόπηση του γεγονότος ότι οι αρχές αυτές είναι κυρίως ρυθμιστικές αλλά διέπουν και τον εποπτικό ρόλο της ΕΣΜΑ σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να τα μελετήσουμε αυτά με προσοχή και να τα αναλύσουμε πριν προχωρήσουμε. Για το ΕΦΡΑΓ και την μείωση του προπολογισμού σε σχέση με το κονδύλι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την έκθεση Μέστατ. Ο νέος κανονισμός για το ΕΦΡΑΓ εγκρίθηκε φέτος τον Ιούνιο και θα τεθεί σε ισχύ την 31η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδο μέσα στη φετινή χρονιά. Κατά την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν χρειάζεται να βεβαιωθούμε από τώρα ότι. Μάλλον πρέπει να βεβαιωθούμε από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ΕΦΕΚΑ έχει τα μέσα για να μπορέσει να φέρει πέρα στι λειτουργίε τη. Η έκθεση μέσα βέβαια προτείνει η ΕΦΡΑΚ να αφήσει κατά μέρο τα πρότυπα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να επικεντρωθεί στις βασικές της αρμοδιότητες. Επίσης, προτείνει ενίσχυση της διακυβέρνησης ε, της έφραξε κατά πολλούς τρόπους, γιατί λόγου χάρη προτείνεται η ΕΦΡΑΓ να αξιολογεί κάθε πτυχή ενός προτύπου και όχι μόνο την τεχνοκρατική του διάσταση. Αυτό με το νέο πρόεδρο της ΕΦΡΑΚ που θα αμείβεται απευθείας από αυτόν τον προπολογισμό και με το συμβούλιο που θα συναντάτε 10 φορές το χρόνο και όχι 4 όπως παλιότερα, αλλάζει τα δεδομένα. Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται και από την ε, κατάλληλη ε, στελέχωση του οργανισμού, αλλά να υπάρχει και απαραίτητη λογοδοσία συμπεριλαμβανομένη τη υποβολή εκθέσεων στην αρμόδια Εθνιστική Επιτροπή προ το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βεβαίω. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει απαραίτητη στελέχωση για να αναλυνθούν και να καλυφθούν αυτές οι νέες αρμοδιότητες. Επίσης υπάρχει και το θέμα των διεθνών σχέσεων που θα έχει και αυτό βεβαίω το δικό του κόστο ω δραστηριότητα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι τομεί δράση όπου θα πρέπει να αναπτυχθεί η ΕΦΡΑΚ. Δηλαδή την δημιουργία δεσμών με τον πανεπιστημιακό χώρο, την τόνωση τη πανεπιστημιακή έρευνα, την πρόθεση της εκπαίδευσης, όχι με την εκπόνηση αυτών καθ' αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά τη στήριξη των εκπαιδευτικών προσπαθειών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η πρόοδος έχει ήδη επιτελεστεί σε σχέση με την ελοποίηση των συστάσεων της έκθεση ΜΕΣΤΑΤ, αλλά παρά τι συστάσεις αυτέ, ώστε να υπάρξει επικέντρωση στι βασικέ αρμοδιότητε τη ΕΦΡΑΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η ΕΦΡΑΚ θα πρέπει να έχει τους απαραίτητου πόρου για να τα φέρνει όλα εις πέρας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα να δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή μας για μια σύντομη απάντηση. ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω δεν θα ήταν πολύ συνετό να σχολιάσω τη συζήτηση στην οποία δεν συμμετείχα, γιατί έπρεπε να παρευρεθώ στη συνεδρίαση και άλλες, ε, σε άλλη επιτροπή. Ευχαριστώ όμως τον κύριο Ντεμπέκερ για την σύντομη εισήγηση που έδωσε εκ μέρους μου. Είναι μια συζήτηση που με ενδιαφέρει προφανώς ιδιαίτερος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε αργότερα αφού συζητήσουμε το επόμενο σημείο, για το οποίο έχουμε περίπου 30 λεπτά το πολύ. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5. Ευρωπαϊκό εξάμεινο για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, υλοποίηση των προτεραιοτήτων για το 2014. Εισηγητή ο Φιλίπ Τεμπάκερ. Σα δίνω το λόγο. Thank you, uh, Chair. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για όσους βρίσκονται εδώ για δεύτερη θητεία να πω ότι ξανά ξεκινάμε. Αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει πολλές φορές παρά το γεγονός ότι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο πολιτικής αυτό το οποίο σχολιάζει μία από τις πιο, τις πιο έντονες συζητήσεις που είχαμε και στο παρελθόν αλλά και τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Σας παρουσίασα λοιπόν την, ε, το σχέδιο έκθεσης το οποίο αφορά διάφορα θέματα τα οποία τα επεξεργάζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε λίγο πολύ να τηρήσουμε την ίδια σειρά επεξεργασία και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε κάνει με τις ομάδες στους προηγούμενους κύκλους που συζητήσαμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δεν θα συζητήσω όλη την έκθεση, την έχετε όλοι, μπορείτε να την διαβάσετε. Θα ήθελα μόνο να ε, σημειώσω κάποια σημεία. Είναι σημαντικό καταρχάς να συνειδητοποιήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια σε καιρούς δύσκολους οικονομικούς το Κοινοβούλιο συμφώνησε με τα κράτη-μέλη να ξεκινήσει μια διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης και νομίζω ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να τηρηθούν παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο για κάποια κράτη-μέλη να του στηρίσουν και να τηρήσουν την ισορροπία του προπολογισμού και να συνεχίσουν την πολιτική λιτότητα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει αυτή η γραμμή και να εφαρμόζεται. Κατά δεύτερον, όπως είπα, αυτή η Συμφωνία Οικονομικής διακυβέρνηση ελήφθη από κοινού με τα κρατημέλη. Στη γνωμοδότηση το διευκρινίζω ιδιαίτερω ότι τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει, ε, θα πρέπει να ξεκινήσουν πλέον να το οικειοποιούνται αυτό το πρόγραμμα για να υπάρξει βελτίωση. Μπορεί μετά από μερικά χρόνια να διαπιστώσουμε ότι είναι μεγάλο το πολιτικό κίνημα, τίμημα mm. και ότι μόνο πάνω από 45% των θεμάτων δεν έχουν καν ε, θυχτεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει ως κοινοβούλιο να το θέσουμε στα κράτη-μέλη. Κατά δεύτερον, μία από τις μεγάλες συζητήσεις που συνεχίζεται σήμερα είναι το θέμα της ε, ανεργίας, κυρίως των νέων. Θα πρέπει να αναφέρουμε λοιπόν συγκεκριμένα το γεγονός ότι θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα και για το Κοινοβούλιο αυτό. Θα ξεκινήσει η συζήτηση. Θα συμφωνήσουμε πολύ ασφαλώ με το πρώτο σκέλο τη διαπίστωση, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται με τη λύση. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει μια εντελογική συζήτηση. Αυτό έγινε και στο παρελθόν. Η δική μου η λύση, όπω αναφέρεται και στην έκθεση, είναι τριών διαστάσεων. Καταρχά, στο πλαίσιο τη οικονομική διακυβέρνηση θα πρέπει να επιμείνουμε για να υπάρχει και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τριορθωτικέ μεταρρυθμίσει και ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Κατά δεύτερον, να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Σήμερα το βλέπουμε ότι ο τραπεζικό τομέα και ο χρηματοπιστωτικό τομέα ακόμα δεν έχουν επανέλθει σε μια φυσιολογική ασφαλή κατάσταση. Να το συνειδητοποιούμε αυτό, να το αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται συνεχής εποπτεία και ανάπτυξη της διακυβέρνηση αυτής και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδοτική σταθερότητα. Ένα παράδειγμα το οποίο συνδέεται και αυτό με την οικονομική ανάπτυξη, ό,τι έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν φτάσει στην ταχύτητα που θα έπρεπε και που ήταν στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερο πυλώνας. Τρίτος πυλώνας. Ο πυλώνας των επενδύσεων ασφαλώς. Ο πυλώνας των επενδύσεων όμως σε ένα ασφαλές πολιτικό πλαίσιο. Όχι μόνο δαπάνη για τη δαπάνη, όχι μόνο χρέωση, αλλά να δαπανάτε τα χρήματα στην ε, έρευνα, την ανάπτυξη, την ε, υγεία, την εκπαίδευση, προκειμένου να αναπτυχθούν όλοι αυτοί οι τομείς και ιδιαιτέρως ό,τι αφορά τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. ιδιαιτέρως ε, με τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί βλέπουμε ότι στον ιδιωτικό τομέα η έλλειψη επενδύσεων αποτρέπει την απαραίτητη ανάπτυξη. Και τελευταίο σημείο, θα έλεγα ότι οι τρεις αυτοί οι πυλώνες από κοινού μπορούν να διαμορφώσουν μια ασφαλή, σταθερή βάση για το πώς ε, θα υποβοηθήσουμε την ανάπτυξη και θα καταπολεμήσουμε την ανεργία στην Ευρώπη. Τελευταίο σημείο και κλείνω εδώ είναι το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας. Βλέπουμε ότι σε όλη τη διαδικασία για την οικονομική διακυβέρνηση υπάρχει έλλειψη οικονομικής, ε, δημοκρατικής συγγνώμη, ευθύνης και λογοδοσίας. Άρα κάνω κάποιες προσπάθειες και κάνω κάποιες προτάσεις για να αυξηθεί η δημοκρατική λογοδοσία. Αυτά τα τρία θέματα λοιπόν ήθελα να θέσω στη συζήτηση. Φυσικά περιλαμβάνονται και άλλα θέματα στη συζήτηση και προσβλέπω στην επικοδομητική συζήτηση με το Κιώδης ε, και με την Επιτροπή Ολόκληρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τώρα οι Σκιώδης Συγητές, Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ο κύριος Ροζάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντα τις ευχαριστίες μου προς τον εισηγητή που συνέταξε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση. Συμμερίζομαι τις περισσότερες από τις απόψεις που ακούστηκαν και όπως προτείνονται στην έκθεση. Να τονίσω τα σημεία που θεωρώ τα πλέον σημαντικά. Το πρώτο έχει να κάνει με την ορθή αποτίμηση τη κατάσταση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωζώνη κυρίω, αλλά και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σωστά δίνεται έμφαση στον ευάλωτο χαρακτήρα τη ανάπτυξη και στου πολλού ε, κινδύνου που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στο μέλλον, για να διασφαλίσουμε την σταθερή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και στο μέλλον. Και ε, σε δεύτερη φάση, κάτι που συμμερίζομαι και στο οποίο πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη προσοχή, είναι το πώ σωστά τονίζει ο εισηγητή την σημασία των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου η Ευρωζώνη να γίνει πιο ανταγωνιστική και να υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Συμμερίζομαι πλήρω τι απόψει του ότι οι διευθυντικέ μεταρρυθμίσει δεν είναι απαραίτητε ω αυτό σκοπό μόνον για τα ενδεχόμενα αποτελέσματα που μπορεί να φέρουν, αλλά μπορεί να εξουδετερώσουν ή τέλο πάντων να αντιμετωπίσουν το κόστο που επιφέρει η δημοσιονομική ενοποίηση. Ε, κάτι, η δημοσιονομική εξυγίανση μάλλον, κάτι που αφορά πολλά κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. Εδώ πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας. Και οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις να υλοποιηθούν βάσει των προγραμμάτων που έχουν προκύψει στις, στις αναχώρας και για τις ε, συστάσεις αυτές καθεαυτές, τις αναχώρα συστάσεις. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επικρίσεις ε, στην έκθεση για το πώς ε, λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός στην Ένεση, ιδίως στην Ευρωζώνη και εδώ θα συμμεριστώ την άποψη του συγκητή. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την υλοποίηση των ε, αναχώρα συστάσεων ευθύς εξ αρχής. Εδώ το περιεχόμενο των συστάσεων είναι ήδη ένα θέμα και ίσως θα μπορούσαμε να καταβάλουμε προσπάθεια να γίνουν πιο ε, ε ισορροπημένες οι συστάσεις αυτές, με πιο μακροπρόθεσμη θεώρηση. Το βασικό πρόβλημα είναι όμως ότι δεν υλοποιούνται εγκαίρως από τι περισσότερες χώρες και η έκθεση προσφέρει και κάποιους, κάποια αριθμητικά στοιχεία. 10% όλων των αναχώρα συστάσεων έχουν υλοποιηθεί, ενώ το 40% έχουν υλοποιηθεί μόνο εν μέρη. Αυτό είναι μια σαφής ένδειξη ότι όλη η διαδικασία δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα με την ανάληψη ευθύνης από τις διάφορε χώρες για τις ε, συγκεκριμένες συστάσεις και την υλοποίησή τους και σωστά υπογραμμίζει ο συγκεκριτής ότι πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους ώστε η εθνική ανάληψη ευθύνη ε, από ε, τα κράτη-μέλη είναι σημαντικό στοιχείο για να λειτουργήσουν και αυτές οι συστάσεις. Κάτι άλλο που βρίσκω σημαντικό και όπου συμφωνώ με τον εισηγητή είναι σε ό,τι αφορά την σημασία των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Ιδίω τι επενδύσει στην εκπαίδευση, έρευνα, ε, ανάπτυξη, καινοτομία, εξοικονόμηση ενέργεια και για τους σκοπούς της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής μας. Στον τομέα αυτό είχαμε τα ισχυρότερα πλήγματα λόγω της ε, οικονομικής κρίσης και βλέπουμε ότι τις προσπάθειες πλέον δεν μπορεί να τις φέρει πέρα μόνο ο δημόσιος λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών. Στους τομείς αυτούς υπήρξε μικρότερη χρηματοδότηση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια και το χαμηλότερο επίπεδο κρατικής, ε, ε, δημόσιας μάλλον ενίσχυσης ήταν ζωτικής σημασίας. Περιορίζεται το δυναμικό και το ποσοστό αποτελεσμάτων και παραγωγής σε όλη την Ευρωζώνη από τους τομείς αυτούς. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι κάτι που το επαναλαμβάνουμε διαρκώς όταν συζητούμε τις μελλοντικές προοπτικές της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η ανάγκη να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά αυτή η ιστορία διαρκώς επανέρχεται. Την αναφέρει και η συγκεκριμένη έκθεση. Αλλά αυτό που προέχει είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει, να εντείνει μάλλον την επιρροή της στα κατημέλη. Επιτέλους να κάνουν αυτά που προκλέπουν οι συνθήκες, να ολοκληρωθεί αυτή η εσωτερική αγορά, ιδίω σε τομεί όπω οι υπηρεσίε, οι χρηματοοικονομικέ και χρηματοποστοτικέ, αλλά και σε άλλου τομεί. Όπω λόγω χάρη πρόσβαση στο κεφάλαιο ή την πηγή χρηματοδότηση για επιχειρήσει. Συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων. Τέλο, ο εισηγητή σωστά υπογραμμίζει τη σημασία τη ε, Μελλοντική Τραπεζική Ένωση και την ανάγκη να δούμε τι θα γίνει με την δημοσιονομική σταθεροποίηση. Ένα εγχείρημα που ακόμη αναμένεται να λειτουργήσει πέραν των ε, μηχανισμών εποπτείας, γιατί τα υπόλοιπα όργανα της Τραπεζικής Ένωσης ακόμη δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί και δημιουργηθεί, αρχίσει να λειτουργούν. Πέραν από αυτών των παρατηρήσεων όμω ε, επί τη έκθεση, έχω και κάποιε ερωτήσει προ τον εισηγητή. Η πρώτη, ίσονο σημασία ζητήματα, αλλά αφήστε με να τα αναφέρω ε, σε κάθε περίπτωση. Το πρώτο, ε, με συγχωρείτε, πρόεδρο. με συγχωρείτε, αλλά έχουμε συγκεκριμένο χρόνο στη διάθεσή μα και έχουμε και άλλου ομιλητέ. Πρέπει να δώσουμε το λόγο σε πολλού συναδέλφου. Ένα λεπτάκι μόνο. Θα με αφήσετε. Ωραία. Για το σημείο 5 προτείνω να μην είμαστε δογματιστές στην προσέγγιση μας. Το κρατικό χρέος βεβαίως δεν δημιουργεί προβλήματα στην ανάπτυξη. Θα έλεγα λοιπόν να μιλάμε για υπερβολική χρέωση και όχι απλώς για χρέος. Ε, επίσης, στο σημείο το, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λογοδοτούν ενώπιον του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των αναχώρα στάσεων Σε κάποιο βαθμό νομίζω ότι αυτό δεν συνάδει πλήρω με τι συνθήκε. Έπειτα το να υπάρχει μια κοινή εκπροσώπηση τη Ευρωζώνη. Με συγχωρεί, Περβάν, σε ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι. Η κοινή εκπροσώπηση είναι σημαντική αρκεί να μπορούμε να μιλούμε με ενιαία φωνή. Εάν αυτό δεν συμβεί, το να υπάρχει απλώ κοινή εκπροσώπηση είναι κάτι θεωρητικό. Είναι σαν να βάζουμε το αμάξι μπροστά από τα άλογα. Θα είμαστε προθύστεροι τρόπον. Επίσης να ενθαρρύνω τον εισηγητή να πει λίγα στοιχεία περισσότερα για το πώς θα βελτιωθεί η διάσταση των ιδιωτικών επενδύσεων. Ευχαριστώ. Thank you for the... Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα Σοσιαλιστές Δημοκράτες Ευχαριστώ. Köszönöm szépen Nagyon fontos jelentés. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση κατά την άποψή μου, διότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στο πλαίσιο της ε, οικονομικής πολιτικής και ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεμπάκερ για τη δουλειά του. Μας ικανοποιεί ιδιαίτερο το γεγονός ότι ο εισηγητής κατάφερε να συμπεριλάβει και να αναφέρει τουλάχιστον κάποιες θετικές αλλαγές σε σύγκριση με τα όσα είδαμε να συμβαίνουν το έτος 2013. Οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες εκφράζουν την ικανοποίησή τους, διότι πολλές από τις βασικές μας προτεραιότητες έχουν συμπεριληφθεί στην πρόταση. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Κατά πολέμηση της ε, φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής, αναφέρονται στο σημείο 24, όπως επίσης η έμφαση που επαναλημμένως δίνεται στην καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας, της ανεργίας των νέων. Θα ήταν σημαντικό επίσης να αναφερθεί καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη και να τονίσουμε και την αρχή της αλληλεγγύης. Μια άλλη θετική αναφορά, ένα άλλο θετικό παράδειγμα στην έκθεση είναι η προάσπιση του δικαιώματος ελεύθερης ε, κυκλοφορίας. Επίσης, η αναφορά στη σημασία της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και η δημοσιονομική εξηγήνση συνοδεύεται από μια άλλη διατύπωση θετική. Βέβαια θα καταθέσουμε και τις τροπολογίες μας, διότι θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε και κάποια από τα συμπεράσματα τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τη προηγούμενη εβδομάδα, τουλάχιστον αυτά με τα οποία είμαστε σύμφωνοι. Επί παραδείγματι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μιλάει για την οικονομική ανάκαμψη η οποία θα υλοποιηθεί όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αν αλλάξουν οι τρέχουσες πρακτικές και πολιτικές της Ένωσης. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε κάτι το οριστικό, τελεσίδου, γιατί όπως και το Φεβρουάριο, έτσι και τώρα θα μπορούσαμε ενδεχομένω ε, να δεχθούμε κάποιους συμβιβασμούς για να έχουμε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Από την άλλη πλευρά βέβαια δεν μπορούμε και να δεχθούμε όταν γίνεται λόγος στην έκθεση για ε, μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν είναι ούτε κοινωνικά βιώσιμες ούτε δίκαιες. Τα όσα αναφέρονται επίσης για την ε, συστάση χώρα. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και αυτή η αρχή φιλική προς την ανάπτυξη, growth friendly. Στο 20 αναφέρεται αυτή η διατύπωση, growth friendly fiscal consolidation. Βέβαια δεν είναι τελείως ε, ορθή διατύπωση σε όλο το σώμα της έκθεσης. Υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις. Εγώ θα πρέπει, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Δεν μπορώ να τα καλύψω όλα, αλλά νομίζω θα βρούμε συμβιβασμού για να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο αυτή την έκθεση. Thank you for the ECR, Mr. Ευχαριστώ πολύ, Τέρχο, για την ομάδα ECR. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ε, διαβάσαμε την έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ. Κατά την άποψή μου εντοπίζει ορθώς ε, τις προκλήσεις. Η ανάλυση της έκθεσης είναι καλή. Υπάρχουν βέβαια και κάποια ε, αποσπάσματα με τα οποία διαφωνώ. σε ό,τι αφορά τα βασικά προβλήματα των ευρωπαϊκών οικονομιών, σωστά αναφέρει ο εισηγητής ότι η έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων εμποδίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Οι δημόσιες επενδύσεις ναι μεν είναι δικαιολογημένες, ενίοτε μακροπρόθεσμα όμως μόνο ο ιδιωτικός τομέας, ένας ισχυρός ανταγωνιστικός ιδιωτικός τομέας μπορεί να βγάλει μια χώρα από την κρίση. Ο εισηγητής αναφέρει επίσης ότι το υπερβολικό χρέος είναι πρόβλημα. Είναι κεντρικό πρόβλημα και ξέρουμε ότι αυτό αποτελεί και ένα άχθος και για τις σημερινές αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Αναφέρει επίσης την ανεργία, την σημασία που έχει ανάπτυξη και θα πρέπει βέβαια να τονίσουμε και ότι η ανάπτυξη εφόσον χρηματοδοτείται μόνο από την κυβέρνηση, δεν μπορεί να είναι ε, κατά ανάγκη βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ανάγκη επίση φοροδιαφυγή φοροαποφυγή είναι σημαντικό. Συμμεριζόμαστε την ε, ε, ανάγκη αυτή. Επίση την ανάγκη για διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει στα κράτη-μέλη. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση για τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξάλληψη των φραγμών για πρόσβαση στην αγορά και πρόσβαση ε, των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Αυτό που δεν τονίζεται στην έκθεση βέβαια είναι η ανάγκη για μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις ομοσπονδιακού τύπου, ο ναι και κάτι σχετικό. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι δίνουμε δεσμευτικές προτάσεις, είναι ένα είδος συμβουλών, συστάσεων. για την οικονομική πολιτική των κρατών μελών. Δηλαδή η Κομισιόν δεν μπορεί να αποφασίζει τι οικονομικέ πολιτικέ των κρατών μελών. Είναι τόσο κεντρική η οικονομία. Αλλά θα πρέπει και οι πολιτικοί να μπορούν να κατανοούν τα πράγματα. Δεν πρέπει βέβαια να επιβάλλονται συστάσεις στα κράτη-μέλη από την Κομισιόν. Η ελευθερία και η δημοκρατία είναι βασικές αρχές. Νομίζω ότι μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξη πολιτική στα εθνικά κράτη να φέρουν σε πέρα στο καθήκον αυτό πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο κ. Παπαδημούλη από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ε, μιλώ εκ μέρου τη ε, ΚΟΕ NGL και τη σκιώδου εισηγητριά μα τη Μαρίζα Ματία, που δυστυχώ λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν μπορεί στη σημερινή μα συνεδρία να είναι παρούσα Λυπάμαι αλλά δεν θα συμμεριστώ τα επενετικά σχόλια για το περιεχόμενο και την κατεύθυνση της έκθεσης γιατί νομίζω ότι εξοραίζει μια πραγματικότητα που είναι ολοφάνερη. Δεν έχουμε μια δημοσιονομική προσαρμογή φιλική προς την ανάπτυξη, αντίθετα έχουμε την Ευρωζώνη μπροστά στο φάσμα μιας νέας ύφεσης. Έχουμε μπροστά μας τον κίνδυνο του αποπληθωρισμού. Πριν δέκα ημέρες μαζεύτηκαν νομπελίστες της οικονομίας όλων των πολιτικών και ιδεολογικών αποχρώσεων και όλοι επέκριναν αυτή την πολιτική που σήμερα κυριαρχεί και επενεί η έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ. Τι φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική προσαρμογή είναι αυτή που στη χώρα μου την Ελλάδα υλοποίησε η Τρόικα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της Κομισιόν και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που έπεσε εντελώς έξω σε όλες τις προβλέψεις. Προέβλεπε συνολική ύφεση 14% και η ύφεση έχει περάσει το 25%. Προέβλεπε το πικ της ανεργίας να φτάσει στο 14% και είναι ήδη στο 30%. Για να μην μιλήσω για την ανεργία των νέων που είναι στο 60%. Και όλα αυτά έγιναν για να γίνει το χρέος βιώσιμο. Και το χρέος πριν αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος ήταν 125% του ΑΕΠ και τώρα έχει περάσει το 175% και πάει προς το 180%. Και το πρόβλημα δεν είναι εθνικό. Το χρέος των χωρών του νότου της Ευρωζώνης είναι μη βιώσιμο και δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη à που έχει κοινό νόμισμα αλλά δεν νοιάζεται να δώσει και μια ευρωπαϊκή απάντηση στο πρόβλημα του χρέους. Είναι γεγονός για να είμαι δίκαιος ότι η έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ κάνει ορισμένες θετικές αναφορές μιλώντας για την ανεργία των νέων που πρέπει να αντιμετωπιστεί και τα λοιπά ή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ή για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Έχετε μελετήσει την πέμπτη έκθεση συνοχής που ετοίμασε η Κομισιόν. Αυτή η έκθεση λέει ότι στα χρόνια της κρίσης από το 9 μέχρι τώρα οι ανισότητες και οι κοινωνικές και οι περιφερειακές αυξήθηκαν. Η φτώχεια αυξήθηκε, η ανεργία αυξήθηκε και η φοροδιαφυγή αυξήθηκε ακόμη και ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Ντράγκη, σε μια από τις τελευταίες του ομιλίες, άσκησε κριτική στην ασκούμενη πολιτική, κομψά, διπλωματικά, όπως συνήθως κάνουν οι τραπεζίτες, αλλά δεν ήταν τόσο υμνητικός και εξοραϊστικός. Είμαστε αντίθετοι με το πνεύμα και τη φιλοσοφία της έκθεσης γιατί η βασική κόκκινη κλωστή που τη διαπερνά είναι ότι όποια προβλήματα υπάρχουν με την ανεργία, με την ύφεση, με τον αποπληθωρισμό οφείλονται στο ότι δεν εφαρμόζεται ακόμη πιο σκληρή πολιτική λιτότητας. Ενώ το ζητούμενο είναι να εγκαταληφθεί αυτή η πολιτική και να έχουμε μια πραγματική στροφή ε, για την ανάπτυξη είναι ολοφάνερο με βάση αυτά ότι δεν συμφωνούμε με την έκθεση ως σύνολο και θα καταθέσουμε στην πορεία για τις δικές μας προτάσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, now for the green. Σας ευχαριστώ για τους πράσινους τώρα. Ο Μπάς Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον Φιλίπ για το σχέδιο έκθεσης. Αυτό που θα κάνω είναι μάλλον να βρω μια μέση οδό μεταξύ αυτών που είπε ο προηγούμενος ομιλητής και αυτά που είπαν οι προηγούμενοι. Γιατί θεωρώ ότι είναι πολλά τα θέματα τα οποία καλωσορίζουμε στην έκθεση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πολλά κρίσιμα ζητήματα όπου διαφέρουν οι απόψεις μας. Και ξεκινάμε με το 1, στο σημείο 1 της έκθεσής σας, όπου αναφέρεται ότι η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι έχει ήδη ξεκινήσει. Λες και πηγαίνουν όλα καλά και θα πάνε όλα καλά στο μέλλον. Ή, εν πάση περιπτώσει, ίσως, Φίλιπ, αυτό να ισχύει αυτό που είπα στην αρχή, ότι Πάμε πάλι από την αρχή. Άλλη μια έκθεση για το εξάμεινο. Χρειαζόμαστε λίγο πιο κατεπήγον χαρακτήρα για την συζήτηση, γιατί δημιουργείται η αίσθηση ότι η έκθεση μας λέει ότι ε, εντάξει, τα χτανίσματα, τα μένουν, ε, κατά βάση βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Όχι. Αυτό θεωρώ ότι θα αποτελούσε λάθος, θα υποτιμούσαμε την κρίση. Ακόμα και ο Ντράγκη το βλέπει αυτό στην παρούσα φάση. Και πιστεύω ότι αν κοιτάξει κανείς ε, τη συνθήκη και την νομοθεσία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιο πολλές από τις συστάσεις αναχώρα, αν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε σε σοβαρή οικονομική ύφεση. Σε αυτή τη φάση λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ περιθώριο στην πολιτική και όχι να συνεχίσουμε business as usual. Άρα να περιμένετε κάποιες ε, τροπολογίες από δική μας πλευράς. Και αυτό μας φέρνει στο επόμενο θέμα. Είπατε ότι θέλετε πιο επί της ουσίας συζητήσεις. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πιο πολύ τη συζήτηση σε ό,τι αφορά τις, εκθέσεις, τις συστάσεις αναχώρα, γιατί η έκθεση είναι σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά γενικόλογη. Λες και έχουν έρθει από ψηλά αυτές οι συστάσεις και δεν μπορούν να τεθούν υπό συζήτηση γιατί οι τρέχουσε συστάσει αναχώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν πολύ σαφή πολιτικό προσανατολισμό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και αυτό θα πρέπει να καταστήσει σαφές και στην έκθεση, γιατί αυτό συζητάμε. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, το κείμενο στο 15 για παράδειγμα, στο σημείο 15 αναφέρεται ότι αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική σύγκληση. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό εξαρτάται από το ποιες ε, συστάσεις συζητάμε. Εγώ μπορώ να αναφέρω κάποιες συγκεκριμένες συστάσεις για τη Γερμανία, για την Ολλανδία, που όντως είναι σημαντικές ε, για την οικονομική σύγκληση, αλλά ακόμα δεν έχουν προκύψει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εδώ πέρα λοιπόν μπορείτε να αναμένετε ε, τροπολογίες. Και περνάμε στο τρίτο θέμα, στη δημοκρατική λογοδοσία. Σημαντικό, γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει και την ε, δημοκρατική λογοδοσία. Το θέτεται μεν το θέμα, αλλά πολύ γενικόλογα προς το παρόν. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και έτσι περνάω στο τέταρτο σημείο, η έκθεση της Τρόικα, την οποία κοιτάξαμε και στην προηγούμενη θητεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό που έκανε με την έκθεση της Τρόικας, ό,τι φορά δηλαδή την άποψη του Κοινοβουλίου, να μας ευχαριστήσει δηλαδή ευγενικά και να την βάλει στο σερτάρι. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τις συστάσεις μας. Πέμπτο σημείο, σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση του πεδίου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, αυτό κάπως λείπει. Αναφέρεται κάποια στοιχεία, μας λείπουν όμως κάποια στοιχεία που είχαν αναφερθεί σε προηγούμενα σε προηγούμενες εκθέσεις Capital Union, Costs, αποτελεσματικότητα των πόρων. Θεωρώ λοιπόν ότι ως βουλευτές δεν θα πρέπει να μείνουμε πίσω και από τους πράσινους θα μπορούσαμε να περιμένουμε αυτή τη διεύρυνση του θέματος του πεδίου και άλλωστε θα μπουν αυτά και στη γνωμοδότηση του, της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Τέλος, αναφέρεστε στην πολιτική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Εγώ που είμαι Ολλανδός, θα ήθελα να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι εδώ. Αν ακούσετε τι γίνεται στις ανακοινώσεις τύπου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε κάποιες χώρες, να μην κατονομιώσω χώρες συγκεκριμένες ε, αλλά η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο είναι μεταξύ αυτών. Ε, μας ενοχλεί λοιπόν το γεγονός ότι δεν είμαστε τόσο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά την πρόληψη της φοροδιαφυγής. Και τώρα στις συστάσεις αναχώρα δεν αναφέρεται αυτή η διάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το διορθώσει αυτό και αυτό θα χαρώ εγώ ιδιαίτερα να το κάνω ως πράσινος και Ολλανδός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπάς λέει ο Πρόεδρος. Η FTD. Έχετε το λόγο. Σα Σας ευχαριστώ και πάλι Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μπάκερ. Είναι δύσκολο να μην συμφωνήσει κανείς. Θέλετε να αυξήσετε την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχουν όντω οικονομικά προβλήματα, οικονομική σταθερότητα, δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο ο τραπεζικό κλάδο και θα πρέπει να γίνονται δαπάνε με σωστό τρόπο. Νόμιζα ότι αυτά τα πήρατε από το μανιφέστο του UKIP. Χαίρομαι λοιπόν που συμφωνούμε από όλων αυτών. Ωστόσο η έκθεσή σα αποτελεί, έχει προβλήματα και στην ανάλυση αλλά και στην πρόταση των λύσεων ε, και σφάλματα οικονομικής φύσεως. Στο σημείο 3 Μιλάτε για την ευρωζώνη και το ότι αυτό καθιστά λιγότερο αμα, ελκυστική την Ευρωζώνη στους επενδυτές αλλά και στους ίδιους και στα ίδια μέλη της Ευρωζώνης ενδεχομένω. Μήπως λείπει αυτό. Κατά δεύτερον, σε ό,τι αφορά την οικονομική σας ανάλυση, αναφέρετε ότι μεγαλύτερος περιορισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το χαμηλό επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων. Η λύση που προτείνεται είναι ακόμα πιο πολύ χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα δημόσια χρήματα. Μα αυτό είναι τμήμα του βασικού προβλήματο μακροοικονομική πολιτική, η οποία δεν συνδέεται με τη χρηματοδοτική πολιτική των εθνικών κρατών μελών. Και εξ αρχή δηλώναμε ότι Μόνο σε επίπεδο εθνικού κρατου μέλη μπορεί κανεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, τα δομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο σημείο λοιπόν, μια πολύ επικίνδυνη πρόταση. Δεν ξέρω αν το προσέξετε στο σημείο 8. Αναφέρεται ότι στη συνάρτηση αυτή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ενιαία εξωτερική εκπροσώπηση της Ευρωζώνης βάσει του άρθρου 138. Αυτό τι σημαίνει το τέλος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κυριαρχίας κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα τα μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αφαιρείτε από τα εθνικά κράτη-μέλη. Αυτός είναι ο σκοπός σας. Αν ναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ. Από τους μη εγγεγραμμένους έχω ένα έτοιμο. Ο κύριος Μονό θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποτίθεται ότι θα καλύπτει, θα μιλτά την οικονομική πολιτική των κρατών, όμως τελικά με το ευρωπαϊκό εξάμεινο καταργείται η εθνική κυριαρχία. Η πατριώτες είναι κατά ε, του, του ομοσπονδιακού κινήματος. Έχουμε ε, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο ως τελευταίο παράδειγμα των καταστροφικών πολιτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την έκθεση του κυρίου Ντεμπάκερ, βλέπουμε ότι απλά ε, επικλήσεις και εξυμνήσεις σε διάφορα γίνονται. Ναι, είμαστε όλοι υπέρ της καταπολέμησης ανεργίας, των διαθοτικών μεταρρυθμίσεων κτλ. Αλλά γιατί να κομίσουμε γλάφκα εσ' Αθήνας. Στο 23 μας λέει τώρα ότι η μετανάστευση δημιουργεί οικονομική ανάπτυξη και θα πρέπει ε, να αξιοποιηθεί. Καμία σχέση δεν υπάρχει όμως μεταξύ των δύο φαινομένων γιατί στη Γαλλία που έχουμε μαζική μετανάστευση δεν θα έπρεπε τότε να είμαστε ε, πρωταθλητές της ανάπτυξης και φυσικά δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση αυτό και γύρω στο 15% των μεταναστών δουλεύουν στη Γαλλία τώρα. Σε ό,τι αφορά ε, τη... τη μείωση των κοινωνικών ε, εισφορών με τον κοινωνικό ΦΠΑ Και αυτή η εξωτερική αντιπροσωπεία, single external representation, τι θα κάνει, θα κάνει τις χώρες κρατήδια, ε, κατά τα γερμανικά κρατήδια. Δεν μπορούμε εμείς να δίνουμε μαθήματα σε χώρες όπως παραδείγματο χάρη είναι η Γαλλία, όταν πάνω από πάνω πολλά δις ε, ράλι δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και όταν βλέπουμε ε, υπερχρέωση σε πολλές χώρες. Thank you. I have now... Ευχαριστούμε. Έχω οκτώ ομιλητές στον κατάλογο. Δέκα. Αλλά θα κλείσω τον κατάλογο των χωριτών με δύο λεπτά ένα ομιλητή. Προτιμάτε να ψηφίσουμε. Εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα και μετά να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία. I ask to prepare the voting cards. Οι συνάδελφοι παρακαλώ να ελέγξουν αν έχουν τις κάρτες τους. Yeah, yeah say we start with the budgetary amendments. Yeah. A test vote first. Test vote. Yes, yes. If everybody is ready, we can test the vote. Εάν είναι όλοι έτοιμοι, όχι λείπει μια, κάποιος δεν έχει την κάρτα του, θα ήθελα να ψηφίσουμε δοκιμαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία δοκιμαστική. Όλοι οι συνάδελφοι παρακαλώ, πέρα τη πληροφορία. Ο κύριος Σίμων δεν έχει κάρτα, πρέπει να τον μετρήσουμε. Άλλοι που έχουν κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Πέρας της ψηφοφορία να ξεκινήσουμε με την πραγματική ψηφοφορία. Πρώτα, Τροπολογίε επί του προπολογισμού. Ξεκινούμε με την τροπολογία 6703 υπέρ, 6723 μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6715 υπέρ, Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Υπεράριθμο το ΕΛΚ. Κατά ένα συνάδελφο. Η μία. Εντάξει τώρα. Πέρας. Απορρίπτεται. 67-25 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67-22 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67-26 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67-06 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67-13. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67-16. Υπέρ. Κατά. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 67-03 έχει υποσχεθει 67-27 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67-07 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 67-28 υπέρ κατά απορρίπτεται 67-04 υπέρ κατά εγκρίνεται 67 όχι, 67, 2, υπέρ, κατά, αποχές, απορριβητέ, 67, 0, 9, υπέρ, 67, κατά εγκρίνεται 67 67.00 υπέρ κατά εγκρίνεται 67.01 υπέρ κατά εγκρίνεται Εγκρίνεται. 67.02 υπέρ κατά Εγκρίνεται. 24. 67-24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αποχές, εντάξει. Αποχές. 67-10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67-17. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67-18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 67-19 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67-21 υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67-12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τα τελευταία δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε. Δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν Στη γνωμοδότηση. 1. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι πρέπει να ελέγξουμε τροπολογία 6 Εγκρίνεται. 26 υπέρ 24 κατά. 7 αποχές. 7 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά. Αποχές Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. απόχέ, Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17, 16 συγγνώμη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. αποχέ. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 με προφορική τροπολογία όχι όχι ε, ξεχωριστή κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές μου φαίνεται ότι απορρίπτεται αποχές Απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά θα ελέγξουμε για την 27 να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική α, με προφορική τροπολογία, πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε προφορικός, υπέρ, κατά,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 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά. Θα ήθελα να ελέγξουμε και την τροπολογία 40. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου όπως τροποποιήθηκε. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 41 υπέρ, 13 κατά, 3 αποχές. Εγκρίθηκε η έκθεση. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα μπορούμε να επιστρέψουμε στην ολοκλήρωση της συζήτησης για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά για κάθε παρέμβαση. Έχουμε δέκα αγορητές. Ο κύριος Μαρίας. Να αναφερθώ σε δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα στα θέματα που έχουν σχέση με την θεσμική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα για τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε μνημόνιο. Αφορά κυρίως σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα. Διότι τι είδους συντονισμός οικονομικών πολιτικών μπορεί να υπάρξει, πώς άλλωστε μπορούν να τηρηθούν οι παρατηρήσεις που κάνει η έκθεση για τις αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο μνημόνιο έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική έχουμε την τρόικα να επιβάλλει τη δικιά της οικονομική πολιτική έχουμε την τρόικα να επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα ζητήματα της φορολογίας και φυσικά όλα αυτά όχι μόνο να μην δίνουν λύσεις στο πρόβλημα του χρέους το οποίο από την ώρα που ήρθε η τρόικα από την ώρα που μπήκαμε στο μνημόνιο το χρέος έφτασε στα ύψη έφτασε στο 178 του αεπ και είναι φυσικά μη βιώσιμο έχουμε αύξηση της ανεργία στο 1,5 εκατομμύριο ανέργους. άρα λοιπόν η πολιτική αυτή έχει αποτύχει και κυρίως όμως η θεσμική υποτίθεται λειτουργία που προσδιορίζει το ευρωπαϊκό εξάμεινο δεν ισχύει. Δεν ισχύει καμιά αρμοδιότητα του ελληνικού κοινοβουλίου, καμιά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τώρα βρίσκονται αυτές τις ημέρες οι υπουργοί της κυβέρνησης στο Παρίσι, διαπραγματεύονται με την Τρόικα και είναι ανίκανοι να επιβάλλουν τα αυτονόητα. Να επιβάλλουν και να ζητήσουν να έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να μειώσει το φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης διότι πέρυσι κρύωσε όλη η Ελλάδα, ξεπάγιασε. Αυτό το απλό ζήτημα που είναι θέμα καθαρά του ελληνικού κοινοβουλίου και το οποίο εγώ πέρυσι εισηγήθηκα ως τροπολογία στην ελληνική βουλή και απορρίφθηκε, απορρίφθηκε με τη λογική ότι δεν προβλέπεται στο μνημόνιο και ότι επιβάλλει η Τρόικα ό,τι θέλει. Επομένως κύριε Πρόεδρε, αυτά που λέμε για θεσμικές λειτουργίες του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση για την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ντελάγκη. Ή η συνάδελφος Ντελάγκη συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Με εγκαταλείπει η φωνή μου σιγά σιγά, οπότε θα είμαι σύντομη και δεν θέλω να ξεκινήσω τη σταδιοδρομία μου σε αυτή την επιτροπή συμφωνώντα με την ομάδα των Πρασίνων. Ε, είναι λίγο δύσκολο, μάλλον επικίνδυνο αυτό που κάνω τώρα. Όχι ακριβώς όπως το προτείνουν οι πράσινοι, αλλά πράγματι την παράγραφο 1 Γνωρίζοντα αυτά που ξέρουμε τώρα, ίσω θα ήταν λίγο αισιόδοξο. Να την ξαναδούμε λοιπόν την παράγραφο 1. Στηρίζω πάντω και συγχαίρω τον εισηγητή Ντεμπάκερ για την έκθεσή του, ιδίω τι σημαντικέ παραγράφου 17, ιδίω για τι συστάσει αναχώρα. Αντίθετα με τον προλαλήσαντα, εγώ θεωρώ ότι οι συστάσει αναχώρα είναι ένα από τα λίγα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων. Και αυτά είναι τα... πρέπει να είναι η βασική μας στόχη αυτή. Όχι γιατί έχουμε φετίχ με τους κανόνες, δεν επιμένουμε γι' αυτό στις συστάσεις σαν χώρα, αλλά πρέπει να, υπάρχει, ε, να υπάρξουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Και ξέρετε, ό,τι και αν συζητήσουμε σήμερα, αύριο μεθαύριο, αν δεν έχουμε διαφορετικέ μεταρρυθμίσει, δεν πρόκειται να πετύχει. Συμφωνώ και στηρίζω λοιπόν ε, τον εισηγητή, αλλά σε ό,τι αφορά το σημείο 24, μια μικρή διαφωνία. Υποστηρίζω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πλουστεύσουν τα φορολογικά του συστήματα, ο εισηγητή. Αυτό με βρίσκει σύμφωνη με χαμηλότερη δασμή για το κόστο εργασία συμφωνώ, αλλά λέει ο εισηγητή, ότι θα πρέπει να έχουμε υψηλότερα δασμού στην κατανάλωση. Η δεν κατάλαβα πού πηγαίνει αυτό. Μιλάμε για τον ΦΠΑ. Δεν έχω καταλάβει, γιατί κάποιοι συντελεστέ είναι τόσο χαμηλοί που δεν μπορούμε να του χαμηλώσουμε ακόμη περισσότερο. Ευχαριστώ. Σωτήρης Ζαριανόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, καταρχήν μια παρατήρηση επί της διαδικασίας η οποία έχει απασχολήσει και την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτέ δεν αποτελούν πολιτική ομάδα. Άρα δεν έχουν εκπρόσωπο και κανεί δεν μπορεί να τοποθετηθεί εκ μέρου του. Το λέω γιατί στην αρχή τη διαδικασία δόθηκε σε κάποιο συνάδελφο ο λόγο ω εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων. Για να τελειώνουμε με αυτό. Όσον αφορά το θέμα μα, παρά τη συνολική διαφωνία του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα με το περιεχόμενο τη έκθεση, πρέπει να πούμε ότι πραγματικά έχει μία πάρα πολύ σημαντική διαπίστωση. Ότι ακόμα κι αν υπάρξει ανάκαμψη από την γενικευμένη και βαθιά καπιταλιστική κρίση, αυτή θα είναι ασταθής, θα είναι ανισόμετρη μεταξύ των χωρών, θα είναι πάρα πολύ ρηχή. Δηλαδή, η ίδια πολιτική η οποία οδήγησε στην κρίση, με την ίδια πολιτική η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να βγει έξω από αυτήν, στηριζόμενοι στο δόγμα το οποίο εκφράστηκε από πολλά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξής φράση «Ευελιξία μεν κάτω από την τρομακτική πίεση των προβλημάτων και των, διαμαρτυριών, αλλά οπωσδήποτε, και αυτό είναι το κυρίαρχο, μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας αυτής που προκάλεσε τα 120 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας, τα 25 εκατομμύρια ανέργους με αυτή την πολιτική οδεύει η ευρωπαϊκή ένωση και το εκφράζει η συγκεκριμένη έκθεση. επικεντρώνει η έκθεση στο ζήτημα της συνέχισης και της ένδεσης των αναδιαρθρώσεων στην αγορά της εργασίας δηλαδή μικρότερη μισθή κατεδάφιση των δημόσιων ασφαλιστικών συστημάτων ιδιωτικοποίηση της υγείας δηλαδή ό,τι αφορά την ε, ζωή του εργαζόμενου του μοναδικού παραγωγού κυριολεκτικά καταστρέφεται. Και μάλιστα καλεί τα κράτη-μέλη να γίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, με συγχωρείτε, να γίνει πολύ πιο αυστηρή προς τα κράτη-μέλη, να υπερβούν τις εσωτερικές διαμαρτυρίες, αντιστάσεις και αντιπολιτεύσεις, ώστε να επιβάλλουν διαπυρός και συνδύρω αυτή την πολιτική. Δίνουν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Τελειώνω παίρνουν κυριολεκτικά από τους και το λόγο και δίνουν στο κεφάλαιο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα. Θα φέρει πολύ περισσότερα εκατομμύρια ανέργους και φτωχούς και ο μοναδικό δρόμο για τους λόγου είναι να ανατρέψουν επί τη ουσία αυτήν εδώ την πολιτική και όσοι την εκφράζουν. Ευχαριστώ. Γκάλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή. Είναι εξαιρετική δομή της έκθεσης. Τρία μόνο σχόλια έχω. Πρώτον, ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς ως πυλώνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλω να τονίσω ότι είναι σημαντικό. Η ενιαία αγορά να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά να μην ε, υπάρξει, να μην υπάρξει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, ορθή εφαρμογή, έπειτα χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να παράσχεται αυτή η υποστήριξη προς τις ΜΜΕ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση. Τρίτον, συστάσει αναχώρα. Συμφωνώ με όλου όσου ανέφεραν τι συστάσει αναχώρα. Πολύ κριτική έχει ακουστεί. Συχνά είναι τεκμηριωμένη και βάσιμη κριτική. Θέλω να τονίσω ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τι εθνικέ κυβερνήσει για, για το περιεχόμενο των συστάσεων αναχώρα, ώστε να πετύχουν αυτέ του στόχου του. Του στόχου που είχαμε προβλέψει όταν εγκρίναμε αυτέ τι τάσει. Θα ήθελα λοιπόν οι παρατηρήσει μου να υιοθετηθούν από τον εισηγητή και να συμπεριληφθούν στην έκθεση. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κυρία Τζιλ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι το σχέδιο της έκθεσης ε, κάνει τη σωστή διάγνωση. Υποδεικνύει ποιες είναι οι αδυναμίες του συστήματος, ποια είναι τα προβλήματα στην Ευρωζώνη. Ανεργία, χρέωση, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, αποπληθωρισμός. Δεν είναι καινούργια όλα αυτά. Ξέρουμε ότι χρειάζεται άμεση δράση και ότι η οικονομία της Ευρωζώνης παραμένει ακόμα αδύναμη. Ξέρουμε ότι δεν ε, λειτουργήσε, δεν λειτουργεί η λιτότητα και ακόμα και ο Μάριο Ντράγκη αναγνώρισε ότι θα πρέπει να τη χαλαρώσουμε. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι τα κράτη-μέλη δεν παίρνουν ε, στα σοβαρά τις συστάσεις χώρα. και ότι αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε ότι κάποιες φορές τα κράτη-μέλη έχουν διάφορους τομείς ε, τους οποίους χρειάζεται να μεταρρυθμίσουν και αυτό δεν αντιμετωπίζεται απαραίτητα με την απαραίτητη διαφοροποίηση, διαφοροποίηση ανακράτης μέλος. Και σε ό,τι αφορά τις διαφορές σε κάθε χώρα αναπεριφέρεια. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να κοιτάξουμε και αυτή τη διάσταση στο μέλλον. Νομίζω ότι θα πρέπει να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει ένα πρόγραμμα επενδύσεων 300 εκατομμυρίων όπως ανέφερε ο Γιούγκερ όπως ε, προανήγγειλε ο Γιούγκερ και αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει ορατό γρήγορα προκειμένου να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη κάποιων Ευρωπαίων πολιτών γιατί στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Νότια Ευρώπη γενικότερα, είναι μεγάλο το βάρος που πέφτει στον πολίτη, βλέποντας το επίπεδο της ανεργίας και το πώς θα βγάζει. Θα πρέπει λοιπόν πραγματικά να χαλαρώσουμε αυτά τα μέτρα λιτότητας και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο αν η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει κάποιες φρέσκες ιδέες, κάποιες προτεραιότητες για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και όχι απαραίτητα να συνεχίσει να ακολουθεί την ίδια οδό, τα ίδια μέτρα. Είναι επιτακτική ανάγκη το, η Ευρωζώνη να βρεθεί στην ίδια, στο ίδιο επίπεδο όπως πολλοί από τους ανταγωνιστές μας, τους εμπορικούς. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, υπερβάνω του περές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την έκθεση του κ. Ντεμπάκερ. Ήθελα να επανέλθω σε ένα-δυο σημεία που θεωρώ σημαντικά. Κατά πρώτον, νομίζω η όλη αυτή προσπάθεια για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, η όλη διαδικασία, στη φάση στην οποία βρισκόμαστε, ως προς την εξέταση εδώ από το Κοινοβούλιο, δείχνει ότι τουλάχιστον στις προτεραιότητες του 2014 να έχουμε επιτύχει πολλά. Βέβαια έχουν αλλάξει και συγκυρίες. Έχει αλλάξει η κατάσταση σε σχέση με τη στιγμή που συλλάβαμε και αρχίσαμε να ελοποιούμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα την κατάσταση. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη όταν συζητούμε την εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Με εντυπωσιάζει λοιπόν, να κοιτάζω την έκθεση του συναδέλφου, σίγουρα είναι μια πρώτη εκδοχή της εκθεσής του και του επιτρέπω φυσικά κάθε είδου δικαίωμα να την μεταβάλει στη συνέχεια αλλά είναι μείζονο σημασία. Δεν μπορούμε να λέμε σε μια τέτοια έκθεση, ε, να μην λέμε μάλλον τίποτα σε μια τέτοια έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σημαίνει ότι τα μέλη της Ευρωζώνης, επειδή είναι σε χειρότερη θέση από τους υπολείπου, δεν μπορούμε να πούμε τι συμβαίνει ακριβώ σήμερα. Ε, έχει υποτιμηθεί το τι συμβαίνει με τις μακρογνωμικές προκλήσεις και την συνολική ζήτηση στην Ευρωζώνη. Αυτά δεν αναφέρονται στην έκθεση. Δεν μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε ότι η ευάλωτη κατάσταση των χωρών της Ευρωζώνης όπως το υπονοεί η έκθεση οφείλεται στις χώρες της Ευρωζώνης που πάντοτε είχαν αξιολόγηση α, αλλά δεν έχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Κάποιοι ίσως να θέλουν να παραμένουν σε αυτό το ιδεολογικό στερεότυπο ή αυτή την προκατάληψη, αλλά καλό θα είμαστε και σοβαροί. Και αν είμαστε σοβαροί, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και να μην ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει κάτι. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει μόνο η οικογένεια των σοσιαλιστών. Το είδαμε και με το IGF όταν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις ίδιες τις, τις προτάσεις. Είδαμε κάποια πράγματα να ε, γίνονται πραγματικότητα. Και οι τελευταίοι αριθμοί μας δείχνουν ότι η ανεργία είναι ανυπόφορα υψηλή, ότι η ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει και ο πληθωρισμός επίσης είναι πάρα πολύ χαμηλά. Εδώ λοιπόν, όσοι μας λένε ότι χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό πρόγραμμα, έχουν κάποιο δίκαιο, αλλά και ε, ο κύριος Ντράγκη που εκφώνησε έναν λόγο τον οποίο σας προσκαλώ να διαβάσετε, δεν ανήκει στην οικογένεια των σοσιαλιστών και λέει ότι πρέπει κάτι να γίνει για τουλάχιστον για τις επενδύσεις. Τίποτα από αυτά δεν αναφέρονται στην έκθεση. Και αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί σε αυτή τη φάση που έχουν φτάσει τα πράγματα, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, υπάρξουν τροπολογίες σχετικά. Ο κύριος Θάλμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή, γιατί πράγματι η έκθεσή του είναι άψογη και πάρα πολύ ισορροπημένη. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Ντεμπάκερ κατά την ε, σύνταξη της έκθεσης την προηγούμενη φορά για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο συγητής ε, ε, τότε και πραγματικά δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ε, οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρηματοδότηση στις ΜΜΕ με βάση τις ανάγκες τους, την κατάστασή τους και όχι μόνο με βάση το που είναι εγκατεστημένες, που έχουν την έδρα τους. Είναι λοιπόν ισορροπημένη, άψογη έκθεση θα ήθελα βέβαια να προσαρμοστεί στις ε, σημερινές τόσο οικονομικές όσο και πολιτικές συνθήκες όπως είπε και η κυρία Περβάν Σουμπερές. Πρέπει να αναφέρουμε και το πρόγραμμα επενδύσεων που πρότεινε ο κύριος Γιούνκερ. Επίσης θα πρέπει να γίνει ε, μια αναφορά γενικώ επενδύσεις. Τίποτε άλλο να στηρίξω τον κύριο Ντεμπάκερ και είμαι στη διάθεσή του να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράιν Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Ντεμπάκρη για την έκθεση του. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη έκθεση και αξίζει να τη λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα να κάνω, να δείξω κάποια σημεία παρ' όλα αυτά. Ποια είναι τα πραγματικά εργαλεία επί των οποίων κρίνουμε μια οικονομία ανεργία, αύξηση ΑΕΠ και στην Ευρωζώνη δεν τα πηγαίνουμε καλά σε σχέση με το με τη ΣΥΠΑ, με τον Εμένα Βασίλειο, είναι διπλάσια ενεργεία στην Ευρωζώνη από ό,τι στη ΣΥΠΑ και στον Εμένα Βασίλειο. Και η ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι λιγότερο από το ίμιση των αντίστοιχων ε, ποσοστών στις ΕΠΑ και στον Εμένα Βασίλειο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο μηχανισμός εποπτείας οι οποίες ε, υπάρχουν θα εφαρμοστούν πλήρω. Λοιπόν, θέλω να πω το εξή. Είναι σημαντική η εποπτεία για όλε τι χώρε, και τι μικρέ και τι μεγάλε. Και τι εννοώ το να καταστούν υπόλογες οι χώρες είναι πραγματικά μία, προοπτική, μία μέθοδος ε, και κινήτρων και φόβητρων. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις ανά χώρα. Ο, ο Υπουργός Σόιμπλε είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Σε μία ομιλία είπε, και να το σκεφτούμε, ότι θα πρέπει να σκεφτούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ως μέσο για να βοηθηθούν οι χώρες με τις ε, συστάσεις αναχώρα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Οι συστάσεις αναχώρα είναι κοστοβόρες, χρονοβόρες, εκφύσεως. Και αν θέλουμε να είναι αποδοτικές όπως όλοι θέλουμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε ο προπολογισμό να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος για να εφαρμοστεί αυτή η σύγκληση των χωρών με τις συστάσεις αναχώρα. Και οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει τα μεγαλύτερα σοκ και η δική μου χώρα έχουν τώρα το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης ΑΕΠ. Και τι μας διδάσκει αυτό, ότι χρειαζόμαστε αντιαθετικές μεταρρυθμίσεις και ότι είναι σημαντικό να κοιτάξουμε το σύστημα της Ευρωζώνης, να υπάρχουν καλά παραδείγματα μεταρρυθμίσεις ε, του δημοσίου τομέα και θα πρέπει να δίνουμε και κίνητρα, όχι να εξαναγκάζουμε. Και τέλος, συμφωνώ με το σημείο της παραγράφου 27 για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 74% τέτοιων, τέτοιες ανάπτυξης στην ΕΠΑ προέρχεται από τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι θέλει ο ιδιωτικό τομέα, βεβαιότητα. Ε, και σήμερα δεν την έχει ακόμα τη βεβαιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα, τελευταίο ομιλητή, Πάτρικ Κοφλίν, και μετά θα δώσουμε το λόγο για τα καταληκτικά σχόλια στον εισηγητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο γινόμαστε μάρτυρε εδώ, στην οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίω τη Ευρωζώνη, είναι διαρκή ενδείξει από τους ε, αντιμάχους της δημιουργίας του κοινού νομίσματος τελικά να επαληθεύονται. Και βλέπουμε να υπάρχει ισοπαίδωση σε τομείς όπως ε, η πρόνοια, η κοινωνική ασφάλιση, η εργασία. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 21. και το διασκεδαστικό. Ενθαρρύνει τα κάτι μέλη να υπερβούν τις εγχώριε πολιτικές διαφωνίε και να εξοχρονίσουν τις οικονομίες τους, την κοινωνική τους προστασία και την υγειονομική πρόνοια. Αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς. Η δημοκρατία. Βεβαίως οι χώρες και τα καθεστώτα που αυτή τη στιγμή ε, ισχύουν θα μπορούσαν να το επιδιώξουν αυτό, αλλά υπάρχουν και οι εθνικές εκλογές. Δεν υπάρχει μηχανισμός που να μπορεί να επιβάλλει τι πολιτικές χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρχει σύγκληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό να ε, είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη. Επίση, κάποιε χώρε που φαίνεται να μην έχουν υπεύθυνη στάση δεν πρέπει να πληρώσουν ε, τα σπασμένα για ευθύνε άλλων. Αυτό που σαφώ χρειάζεται είναι κάποια απόφαση για το πώ θα λειτουργούν τα εργαλεία αυτά σε ευρωπαϊκό ή σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να λειτουργήσει κάτι τέτοιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο μόνο τρόπο να προχωρήσουμε είναι να επανέλθουμε στο εθνικό επίπεδο, κατά την άποψή μα. Και μου κάνει εντύπωση που πολλέ χώρε τη Ευρωζώνη, ιδίω στο νότο τη Ευρώπη, έχουν τελείω διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τη Γερμανία, η οποία διαθέτει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, ερευνά, ε, εμπειρία βιομηχανική πορεία ως τώρα, οι χώρες αυτές θα πρέπει να μπορούν να, το, να, δώσουν, να προωθήσουν το δικό τους νόμισμα και τις δικές τους αξίες με το δικό τους εθνικό νόμισμα. Βάζει τη δική τους οικονομική δραστηριότητα. Πολλοί έκαναν σχόλια για την πρώτη παράγραφο και την ε, ανάκαμψη που μπορεί να έρθει. Νομίζω με τα πρόσφατα δεδομένα θα πρέπει ο συντάκτης να το, να το αναδιατυπώσει στο σημείο αυτό. Δεν θα υπάρξει καμία ανάκαμψη, ιδίω αν τα πράγματα παραμένουν όσο έχουμε το ευρώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατά πρώτον, να πω ότι ότι είμαι επιστήμον και ότι τα θέματα αυτά με έχουν αποσχολήσει από πολλά χρόνια. Προσπάθησα να καλύψω λοιπόν αυτές τις διαστάσεις που αφορούν τους συναδέλφους που του απασχόλησαν στην έκθεσή μου. Φυσικά και υπάρχουν σημεία που λείπουν και αν κάπου χρειάζεται μεγαλύτερη επίπεδο λεπτομέρειας να το συζητήσουμε με τους κοιόδη και να τα ε, αποσαφηνίσουμε. Δεν θέλω όμως να γραφτεί μια 20 σέλιδη έκθεση που να περιλαμβάνει τα πάντα σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο για να ακουστεί ό,τι ε, περνάει από το μυαλό του καθενός. Υπάρξουν, υπήρξαν και κάποιες παρατηρήσεις θετικές, αλλά και κάποια σχόλια από πλευράς μου, ίσως και είδη σύντομων απαντήσεων. Και θα τα ξαναδούμε και στο μέλλον όταν συζητήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις στην Επιτροπή μας. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα είναι αυτό των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων και το αν είναι υπερβολική ή λίγη η λιτότητα, εάν χρειάζεται ή όχι περαιτέρω δημοσιονομική ένωση. Ε, πολλοί θα πρέπει να εξορθολογήσουν ε, την αγορά εργασία του, τα μέτρα που έχουν λάβει και το καθεξή. Αν δούμε την πρόσφατη ομιλία του κ. Ντράγκη, όχι μόνο την ε, πιο πρόσφατη, αλλά των τελευταίων διμήνων όλε του τι παρεμβάσει, ε, καταλήγουμε νομίζω στο εξή συμπέρασμα. Δεν υπάρχουν δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την κρίση στην Ευρωζώνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο με κονδύλια και διοχετεύοντας χρήμα. Είναι θέμα ε, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να αναλάβουν ε, τι ευθύνε του, να κάνουν τι σοβαρές διευθυντικέ μεταρρυθμίσει και η Ευρωζώνη να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανοιχτότερη και να στραφεί περισσότερο προ το εμπόριο και τι εμπορικέ συναλλαγέ. Αυτή είναι η πολιτική μα ευθύνη. Όλοι σε αυτό το κοινοβούλιο ε, νομίζω καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι τεράστια ευθύνη για τι μελλοντικέ γενναίε τη Υπήρου μα. Αυτό είναι η ουσία τη εκθεσή μου και αυτό θα ήθελα να παραμένει και ο κεντρικό τη άξονα και ευχαριστώ για τη στήριξη που δείχνατε προ αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίω τίθεται και το ερώτημα πώ, όπω είπε και ο Μπάς από του πράσινου, πώ με τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία που έφτασαν στα χέρια μα, η έκθεση ήδη την προσφορά τον Ιούλιο, οπότε τα στοιχεία αυτή τη εβδομάδα δεν προλάβαμε να τα λάβουμε υπόψη, θα γίνουν κάποιε σχετικέ μετατροπέ, αλλά και κάποια στοιχεία τη έκθεση Draghi μπορεί να καλύπτονται στην επόμενη εκδοχή της έκθεσης. Υπάρχουν και άλλες επίσης πρόσφατες δημοσίευσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη, αλλά δεν υπάρχει λόγος, ε, εφόσον αναφέρουμε τις εκθέσεις αυτές και γίνονται οι σχετικές να πηγαίνουμε στις λεπτομέρειές τους και στα συμπεράσματά τους και να τα αναφέρουμε και αυτά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Ε, υπήρξαν πάρα πολλές άλλες παρατηρήσεις, αλλά θα περιμένω περισσότερο την επόμενη συζήτηση, δεν θα περάσω τώρα σε λεπτομέρειες, διότι νομίζω ότι ήμουν σαφή. Νομίζω ότι υπάρχει ε, στήριξη από πολλές διαφορετικές ομάδες προς αυτή την κεντρική κατεύθυνση, αλλά βεβαίως οι παρατηρήσεις που αφορούν τις λεπτομέρειες θα ληφθούν υπόψη στη συνέχεια. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε από κοινού να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσω το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες προθεσμία. Έχει οριστεί 8 Σεπτεμβρίου 12 το βράδυ, λέει ο δώσαμε μία μικρή αναβολή μέχρι τα μεσάνυχτα για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρον το χρόνο μας, γιατί έχουμε και θέματα μετάφρασης. Θα γίνει η συζήτηση 22 και 23 Σεπτεμβρίου, 7 Οκτωβρίου ψηφοφορία στην Οίκον και στην Ολομέλεια στην δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο στις 9 με τον πρόεδρο του Ευρωγκρουπ, τον κύριο για τον οικονομικό διάλογο.